αλλά που είναι μια ένωση πολιτική και στο τέλος μπορούμε να την αποκαλέσουμε και ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ κυρία Κόμη. Πέρα τη συζητήσεως, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τώρα στην ημερήσια διάταξή μας έχουμε την έκθεση Ακούνιε που αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών. Δίνω παρευθύ το λόγο για ένα τετράλεπτο στην εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το κείμενο είναι σημαντικό διότι οι δύο στόχοι είναι να έχουμε σταδιακή και αρμονική ανάπτυξη του συστήματος ηχτονική αναγνώρισης των βοηδών με μια ρήτρα αναθεώρησης σε πέντε χρόνια για ενδεχόμενο πέρασμα σε ηλεκτρονική αναγνώριση υποχρεωτική. Το δεύτερο σημείο που εμπεριέχεται και είναι σημαντικό στον κανονισμό είναι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την προσθήκη της αναφοράς της δυνητικής ευχέρειας που υπάρχει όσον αφορά την αναφορά που θα υπάρχει στα πακέτα με το, βοη... με με το βόλιο κρέας. Ε, περνάμε από την Ολομέλεια τώρα για να διορθώσουμε τις ασυνέπειες που υπήρχαν όταν ψηφίσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Υπήρξε ε, κάποιο πρόβλημα από πλευρά των υπηρεσιών τη ε, Επιτροπή μετά από διαβουλεύσει με ειδικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνω το εξή. Σήμερα να εγκρίνουμε τρει τροποποίησει που έχουν αποκλειστικό στόχο τη διόρθωση των ασυνεπιών και τη διευκρίνηση του κειμένου. Οι τροπολογίες μου 45 και 47 αποτελούν απλώς τεχνικές διορθώσεις. Η τροπολογία 46 προτείνει ότι απλούστευση της διαδικασίας της δυνητικής ετικετοθεσίας να μην τεθεί σε ισχύ παρά πρωτη η του 2014 και υπενθυμίζω ότι αυτή η αναφορά, η δυνητική, θα πρέπει να είναι αντικειμενική, αληθής, επαληθεύσιμη μάλλον από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητή για τον καταναλωτή. Για να αποφευθεί κάθε αβάσιμος φόβος εδώ. Επίσης επαναδιευκρίνησα ότι η αρμόδια αρχή επαληθεύει την αλήθεια των αναφορών που τίθενται εθελοντικά και στο 22 παράγραφος 4α προτείνονται κυρώσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε αντίθετη περίπτωση. Εδώ αναφερόμαστε σε ε, κάτι που γίνεται εθελοντικά και όχι υποχρεωτικά και είναι κάτι που αφορά την αναφορά προέλευσης του κρέατος. Μιλάμε για εμπορική πληροφορία που χρησιμοποιείται από τους εμπορευομένους όταν θέλουμε να προστευτούν οι κανόνες για το πιο, πιο ξεκάθαρα. Όσον αφορά λοιπόν την ηλεκτρονική αυτή αναγνώριση των βοηδών, συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών. Δεν είμαι υπέρ της ιδέας περιορισμού του γεωργικού αυτού τομέα, δηλαδή υποχρεωτικά άμεσα να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Είμαι νομοθέτης και φρονώ ότι είμαστε υπεύθυνοι σήμερα για τους νόμους που ψηφίζουμε που έχουν οικονομική συνέπεια. Ο τομέας του, βοηδό, του βοηού κρέατος στην Ευρώπη, στην Ευρώπη και του, των βοηδών υποφέρουν σήμερα. Υποφέρουν και δεν μπορούμε εμείς οι νομοθέτες να τους υποχρεώσουμε να δαπανίσουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα δημοσιογείας που τίθεται εδώ, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης για καλύτερα ανιχνευσιμότητα των βοηδών που θα επιβληθεί με την πάω του χρόνου στον τομέα και θα δούμε σε πέντε χρόνια αν πράγματι είναι ασφαλής η τεχνολογία και αν ο τομέας ή οι τομείς είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν και ίσως η οικονομική συγκυρία να είναι τότε καλύτερη. Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα, δηλαδή την ετικετοθεσία των βοηδών, περί τίνος πρόκειται. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ετικετοθεσία, την εθελοντική. Δεν ε, το καταργούμε αυτό. Θέλουμε να απλουστεύσουμε το σύστημα, να απλουστεύσουμε τη διαδικασία. Εξηγούμε απλούστατα. Η ετικετοθεσία των, του κρέατος αφορά όλα τα είδη κρέατος, με το ίδιο τρόπο εφαρμόζεται. Για το βόλιο κρέας η διαδικασία περιεπλάκει λόγω της ασθένειας των τρελών αγελάδων. Εγώ τι λέω, ας κρατήσουμε τη δυνητική ευχαίρεια, την ε, θελοντική εφαρμογή, απλουστεύοντας όμως το σύστημα, διότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς για αυτό το διοικητικό άχθος, το οποίο σαρκώνουμε εμείς στις διαδικασίες μας. Και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προστεύσουμε τις διαδικασίες υπέρ των πολιτών μας. Αυτά και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει η Επίτροπος, η κυρία Ρέντιν. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευγνωμονεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που προσέφερε σε αυτή την πρόταση για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοηδών και για την απλούστευση της ε, ετικετοθεσίας για το βόηο κρέας και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, την κυρία Οκονή, ε, για την δέσμευση που έχει επιδείξει. Ελπίζω ότι η αφοσίωσή της πραγματικά θα οδηγήσει σε υιοθέτηση του κειμένου σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό θα είναι εξαιρετικά καλό, διότι ε, οι κανόνες που προτείνονται είναι μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί ο κλάδος και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις. Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο ε, σύστημα ανιχνεσιμότητας είναι αποτελεσματικό για την προστασία του καταναλωτή. Η ηλεκτρονική όμως ταυτοποίηση θα ε, κάνει το σύστημα πιο γρήγορο, θα βελτιώσει ε, ε, τις λειτουργίες και θα έχουμε ε, καλύτερη διαχείριση κάθε, του προβλήματος κάθε φορά που ξεσπάει μια ασθένεια και θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα σε γενικότερο πλαίσιο. Απλουστεύονται οι διαδικασίες, αξιοποιούνται ε, οι νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι η σύγχρονη τεχνολογία απέχει μόνο ένα κλικ από τον Ευρωπαίο αγρότη και είναι καθήκον μας να υιοθετήσουμε νομοθεσία έτσι ώστε να αξιοποιήσει ο Ευρωπαίος αγρότης όλες αυτές τις δυνατότητες. Ως προς την το έχει ήδη ε, καταρτιστεί οριζόντια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το βόλιο κρέα καλύπτεται με τον ίδιο τρόπο όπω οποιαδήποτε άλλο κρέα, άρα δεν ε, υφίσταται καμία ανάγκη να έχουμε ειδική διαδικασία έγκριση. Οι φορεί εκμετάλλευση, οι επιχειρήσει τηρούν τι οριζόντιε διατάξει και αν το κάνουν αυτό μπορούν βεβαίως να προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίε όμως δεν θα πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή και θα πρέπει ε, να αναθεωρηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Να έχουμε υπόψη μας και την υφιστάμενη νομοθεσία για την εθελούσια ετικετοθεσία του βόλιου κρέατος και για το γεγονός ότι αυτή έχει χαρακτηριστεί ως πολύ επαχθής για την βιομηχανία έχει χαρακτηριστεί έτσι στο αντίστοιχο κείμενο της Επιτροπής ε, το οποίο αναφέρεται στη μείωση ε, του φόρτου και της γραφειοκρατίας που θα πρέπει να φέρουν σε πέρας οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερος και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο διότι κινείται ε, προς τη δική μας κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Συνάδελφε Γκέρλινγκ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό για την Επιτροπή Γεωργίας. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο κύριος Νίκολσον, ο οποίος είναι ο εισηγητής ε, ε, για την Επιτροπή μας, ε, καθυστέρησε ερχόμενος εδώ. Θα έρθει σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, λοιπόν, εσάς και τις υπηρεσίες. Απλά να πω πως εγώ εκφωνώ τον λόγο του συναδέλφου. Θα ήθελα λοιπόν να παρέμβω λόγω της πρόσφατής μου εμπειρίας με την ηλεκτρονική αναγνώριση, αναγνώριση στα πρόβατα. Το σύστημα αυτό επιβλήθηκε στους αγρότες στην περιφερειά μου παρά την αντίστασή τους και τώρα υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό και ξέρουμε πως δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Δεν σημαίνει αυτό πως δεν το βρίσκουν χρήσιμο κάποιοι αγρότες, ειδικά εάν θέλουν να διαχειριστούν το κοπάδι τους, αλλά δεν μπορεί να είναι το κύριο σύστημα για την παρακολούθηση των ε, μετακινήσεων των κοπαδιών. Και αυτό φαίνεται από το ότι, παραδείγματο χάρη, η Κομισιόν έδωσε περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εφαρμόσει το σύστημα. Γιατί να επεκτείνουμε το σύστημα στα βοηθή πριν ε, λύσουμε τα προβλήματα που έχει και γιατί να το επεκτείνουμε ούτω ή άλλω ε, χωρί να είμαστε σίγουροι για τα ωφέλη. Εδώ πέρα μιλάω βέβαια για την υποχρεωτική βάση του. Τρομοκρατούνται οι αγρότε για το ότι δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την πολλαπλή συμμόρφωση και άρα δεν θα λάβουν τι επιδοτήσει του. Θα πρέπει λοιπόν να εργάζονται εξυπνότερα οι αγρότες και οι αρχές. Αυτό πρέπει λοιπόν να κάνουμε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Εν ονόμα των πολιτικών ομάδων μου, αγορητέ, Για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Και... Συνάδελφε Λίζε, απουσιάζει. Συνάδελφος Λίζε. Αντικαθίσταται από τον συνάδελφο Αγιούζο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε να, να ευχαριστήσω εσάς αλλά να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, την κυρία Οκονή για τη δουλειά της. Καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό. Συμφωνώ απολύτως με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως προς την ταυτοποίηση, την ηλεκτρονική ε, ταυτοποίηση του βόλου κρέατος. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω το ίδιο ως προς το σύστημα της εθελούσιας ετικετοθυσίας για το βόλιο κρέας. Η πρόταση κατάργησης ε, του, που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ούτε είναι και η καλύτερη. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι κερδίσαμε πάλι την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου καταναλωτή ε, για το, στο βόλιο κρέας. Στα επιχειρημάτα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπογραμμίζεται το υποτιθέμενο διοικητικό άχθος. Ενώ αυτό δεν ισχύει, γιατί όλα αυτά τα διαδικαστικά τα γνωρίζουν απόλυτα και πολύ καλά οι δημόσιες αρχές. Για παράδειγμα, στη χώρα μου έχουν εγκριθεί 180 ε, τέτοιου είδους ετικέτες για βόλιο κρέας αλλά μόνο 32 για ε, ε, κατσικίσιο ή για κρέας άλλης προέλευσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα εργαλεία είναι πολύ ε, αξιόπιστα και πολύ χρήσιμα. Ο καταναλωτής θέλει να ξέρει τι αγοράζει και τι καταναλώνει. Δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της εθελούσιας και της υποχρεωτικής ετικέτας. Και πολύ συχνά ε, ο καταναλωτής θεωρεί ότι είναι πιο σημαντική η εθελοντική ετικετοθεσία, μια ετικέτα που έχει μπει σε εθελούσια βάση παρά η υποχρεωτική και δίνει πολύ περισσότερη σημασία σε αυτό. Δεν λέω ότι ο κανονισμός 1770 του 2000 είναι τέλειος, αλλά είναι καλύτερο από τον, αυτό που προτείνεται. Αν καταργηθούν τα άρθρα 16, 17 και 18 θα έχουμε ένα ε, νέο σύστημα χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικός εξωτερικός έλεγχος. Προτείνουμε λοιπόν να ε, εδρεωθούν συγκεκριμένοι ε, κανόνες ανακλάδο για το συγκεκριμένο κλάδο του βόηου κρέατος. Αυτό υπάρχει ήδη σε άλλους τομείς, στον τομέα των πουλερικών για παράδειγμα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο ήδη το εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος θέλω να πω ότι η ετικετοθεσία πραγματικά είναι καθοριστική ε, τη στιγμή που κάνει ο καταναλωτής, ο επιλογέ τις επιλογές του. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνουμε πολύ εξημών ε, στην Ολομέλεια εδώ γιατί ε, τώρα θέλουμε να αλλάξουμε ένα σύστημα που έχει λειτουργήσει τόσο ικανοποιητικά όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για σας και Δημοκράτες, κύριε κυρία Ροθπέρεν έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα, όταν πριν από 15 χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης της ε, σπογκόδους ε, κεφαλοπάθειας που ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής, εάν φοβόμουν τόσο, τότε δεν θα είχαμε σήμερα την ασφάλεια του βοδινού κρέατος στην οποία σήμερα μπορούμε να βασιστούμε. Πριν από 15 χρόνια ήταν αυτονόητο ότι θα υπάρξει διαβατήριο των ζώων και θα είναι υποχρεωτικά δύο ενότια στα αυτιά του ζώου. Και σήμερα καθυστερούμε. Δηλαδή χρειάζονται κρίσεις για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Η εισηγήτρια είπε πως μιλάμε ε, πως δεν μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Κι όμως, ακριβώς γι' αυτό μιλάμε. Για τη δημόσια υγεία, αυτό είναι το θέμα. Και παραδέχομαι πως βεβαίως η εισαγωγή ενός υποχρεωτικού ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης σημαίνει κόπο και έξοδα. Γι' αυτό εγώ πρότεινα στην Επιτροπή να δώσουμε μια μεταβατική περίοδο 10 ετών. 10 ετών αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά ούτε και αυτό δεν μπόρεσε να δεχτεί η πλειοψηφία της Επιτροπής. Δηλαδή θέτε να πάτε σοβαρά στους ψηφοφόρους σας και να τους πείτε πως μιλάτε σοβαρά για τη δημόσια υγεία με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποιος αγρότης θα έλεγε δεν μου φτάνουν 10 χρόνια. Και μετά για την σήμανση. Πάντα λέμε πως ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να έρθουν πιο κοντά στον καταναλωτή, να δώσουν πληροφορίες που τους ενδιαφέρει. Ποια είναι η ηλικία των ζώων, πώς έζησαν, με τι τράφηκαν ε, κτλ. Αυτή τη δυνατότητα έχουμε με αυτό το εθελοντικό σύστημα και χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα προτείνει η εισηγήτρια τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά να διαγραφούν με τους όρους που έχουν. Δηλαδή θα, έχει ένα σύστημα το οποίο θα, θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει όρους. Ε, πώς θα λειτουργήσει. Καμία εθνική αρχή δεν θα είναι σε θέση να ελέγξει οτιδήποτε. Ε, δεν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλει να διαταράξει και το υφιστάμενο σύστημα. Ευτυχώς η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατηρήσει το εθελοντικό σύστημα ως έχει και παρακαλώ τους συναδέλφους να στηρίξουν τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην αυριανή ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης θεωρώ πως πρέπει να σκεφτούμε την διοικητική απλοποίηση του συστήματος, αλλά να απλοποιήσουμε το σύστημα και τη διοικητική του πτυχή. Να βοηθήσουμε τις αρχές. Αλλά αυτό το οποίο προτείνεται εδώ πέρα είναι λανθασμένη προσέγγιση. Παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε και το συμφέρον των καταναλωτών και των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για την Άντε έχετε το λόγο συνάδελφε Μάνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Οκόνη. Ήταν έξοχη δουλειά που έκανε. Το θέμα είναι πολύ τεχνικό, αλλά συζητήτε. Η ασφάλεια των τροφίμων σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, επουδενή, δεν θέλουμε εκ νέου να γνωρίσουμε την κατάσταση που γνωρίσαμε δεκαετία του 90 με την κρίση της τελής Αγελάδας. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα ζώα. Κάθε εκμετάλλευση, κάθε ζώο θα πρέπει να είναι καταχωρημένα. Η παρακολούθηση των ζώων θα πρέπει ε, να εφαρμόζεται δεν ελήφθη υπόψη η τεχνική αναγνώριση, η ηλεκτρονική αναγνώριση στην παρούσα νομοθεσία. Απλώς τα ενότια προβλέπονται. Ε, είχα, σε επαφή με πολλούς παραγωγούς όσον αφορά το σύστημα και πώς λειτουργεί το παρόν με τα ενότια. Ε, προχώρησε η τεχνολογία και ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι τα μέσα ηλεκτρονικής αναγνώρισης ε, έχουν εξυγχρονιστεί. Έκανε σημαντικό βήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι για τη θέση που πήρε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και χαίρομαι προχωρούν προσεκτικά. Ε, η χρήση αυτής της αναγνώρισης ε, θα γίνεται επεθελουσίας ε, βάσος για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα δοκιμαστεί ήσυχα θα πρέπει να είναι θελοντικό το σύστημα επίση που εφαρμόζεται την δικαιοθεσία του βοήου κρέατο. Υπήρξαν πολλά κενά στο παρόν σύστημα και υπάρχουν πολλέ διαφορέ από κράτο σε κράτο. Κάποια κράτη-μέλη δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το σύστημα και γι' αυτό θα πρέπει το σύστημα να είναι σαφέστερο ώστε οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους τις καλές πληροφορίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ECR, ο κύριος Βοητσεκόφσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η ομάδα ECR υποστηρίζει την έκθεση, συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Είμαστε υπέρ ηλεκτρονικού συστήματος αναγνωρίσεως των ζώων να εφαρμόζεται θελοντικά το σύστημα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος είναι δύσκολη και κυρίως είναι δαπανηρή και μάλιστα για τους μικρότερους παραγωγούς, τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις οπότε θα πρέπει να εφαρμόζεται εθελοντικά και είναι σημαντικό αυτό Όσον αφορά την ετικετοθεσία του βοήου κρέατος, πρέπει να υπογραμμίσω μια σημαντική τροπολογία που αφορά την αναγκαιότητα τη ετικιοθεσία όσον αφορά το κλωνοποιημένο κρέα ή μάλλον το κρέα που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα. Είναι περιθωριακή σημασία σε αυτή τη φάση αλλά αν αυτό, αυτού του είδους το κρέας χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αναφέρεται, να εντοπίζεται. Ρώση, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση οδηγία, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, εάν δεν αλλάξει πολύ από ε, θα μα βρει αντιθέτω. Από τη μια πλευρά έχετε, δίνει τη δυνατότητα στου χνοτρόφους να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική αναγνώριση και είναι πιο αξιόπιστα τα στοιχεία έτσι. Και είναι μεγαλύτερη χρησιμότητα και ασφάλεια των τροφίμων και αυτό εφαρμόζεται θελοντική βάσεω. Απ' την άλλη όμω θέλει να απαγορευτεί η ετικετασία θελοντική. Θεωρούμε να είναι παράλογο να μην μπορεί να αναφέρονται στην ετικέτα συμπληρωματικέ πληροφορίε ε, Όπω είναι η ράτσα ή το φύλλο του ζώου, η τροφή που χρησιμοποιήθηκε, το ηλικία του ζώου, οι άλλε ενδείξει που θα μπορούσαν καθαρά να ε, ξεχωρίζουν το ένα είδο βοήου κρέα από το άλλο. Γιατί θέλει να καταργήσει ένα σύστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου εφαρμόζεται εθελοντικά με τη δικαιολογία ότι δημιουργείται ένα μεγάλο διοικητικό άκθος. Ο καθένας όμως κτηνοτρόφος μπορεί να αποφασίσει εθελοντικά να το αναλάβει θα μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτή τη μεθοδολογία. Πιστεύουμε ότι αν, υπάρχει αυτή δυνα... αν δεν υπάρχει δυνατότητα, ε, δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και έτσι δεν δίνονται πληροφορίε στους καταναλωτές. Ευχαριστώ για τι μία εγγεγραμμένου. Συνάδελφε Γκρίφιν, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το εθελούσιο σύστημα πράγματι θα επηρεάσει το βρετανικό. Ε, αν και το Βρετανικό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί ψηφοφόροι μου έχουν πει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μεταφορά των ζώων των ζώων μπορεί να ε, τελικά να διευκολύνει τη μεταφορά των ζώων για σφαγή. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου απαραίτητο ε, σήμερα που έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες ψήξης. Δεν είναι απαραίτητο η διάνυση πολλών χιλιόμετρων για όλο αυτό ε, το πράγμα το κρέας που προέρχεται από ε, ζώα τα οποία υποφέρουν ε, τη σφαγή με βάση θρησκευτικό το λειτουργικό ε, θα πρέπει να επισημαίνεται για να μπορούν να το απορρίψουν οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στους άλλους αγορητές ο λόγος τώρα. Συνάδελφε Σνέλχαρτ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήδη υπόθηκε πως πριν από πολλά χρόνια στην κρίση της φογκώδης κεφαλοπάθειας λάβαμε μέτρα και υποχρεωτικά και εθελοντικά που οδήγησαν στο να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καναλτών στο βόηο κρέας. Και νομίζω πως Νομίζω πως ένα τέτοιο σύστημα οδήγησε και σε ανταγωνισμό στην αγορά. Μιλάω για τα εθελοντικά στοιχεία τα οποία δεν θέλουν να χάσουν κάποιοι ως ένδειξη και τώρα μιλάμε για διαγραφή τους. Βεβαίως να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και η συγγήτρια έχει υποβάλει μια πρόταση για το πώς ε, ακριβώς ε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Το άρθρο 7 απαγορεύει ε, παραδείγματο χάρη διάφορα πράγματα. Αλλά ερωτώ την Κομισιόν, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους ε, από πλευράς ε, κομισιών ή επαφίονται όλα στα ε, κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα του νέου συστήματος όσον αφορά δε τη σήμανση της προέλευσης των ζώων. Εδώ πέρα χρειάζεται νομίζω θάρρος. Όταν λέμε πως δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει πρώτα απ' όλα να εισαχθεί, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά να υπάρχουν και δύο συστήματα σε μια εσωτερική αγορά δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται ένα σύστημα για το εμπόριο και αυτό μπορεί να είναι μόνο ηλεκτρονικό. Όταν παραπονιούνται ε, πως ε, τιμωρούνται οι αγρότες όταν λείπει το ένα ενότιο και χάνουν τα λεφτά λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς αυτό θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Αρσένη έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με λύπη μου είδα για ακόμη μια φορά στο κοινοβούλιο αυτό και αυτή τη φορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να καταψηφίζεται μια τροπολογία για τη σήμανση των ε, προϊόντων βοηδών ε, που διατρέφονται μεταλλαγμένα. Αναρωτιέμαι ποιος δεν θέλει οι πολίτες να γνωρίζουν τι καταναλώνουν, ποιος δεν θέλει οι πολίτες να επιλέγουν και ποιος υποστηρίζει τα συμφέροντα των εταιριών ή αυτό που νομίζουν οι εταιρείες ότι τους συμφέρουν να λειτουργούν κρυπτό. Αντίστοιχα ε, και στα θέματα της χνηλασιμότητας. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που μπορεί να γλιτώσουμε αν έχουμε τη σωστή χνηλασιμότητα και με την ηλεκτρονική σήμανση μπορεί να, έχουμε, να γλιτώσουμε πραγματικά θανάτους, απώλεια ζώων συμπολιτών μας από ε, αρρώστες και επιδημίες. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια εκ μέρου των Σοσιαλιστών, την κυρία Ντάγμα Ρουθ Μπέρετ, για την εξαιρετική δουλειά τη. Ελπίζω η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να ανατρέψει ε, κακά αποτελέσματα στην Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, και να λειτουργήσει πραγματικά προστατευτικά στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Ράιμερς, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, θεωρώ πως ε, πρέπει εδώ πέρα να προσέξουμε για το ότι μιλάμε για δύο θέματα. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στην εθελοντική σήμαση των βοηθών, αλλά στην ηλεκτρονική σήμαση των ζώων. Και εδώ πέρα, κύριε Σνελχάρτ, πρέπει να αντιταχθώ. Όσοι τρέφουν εγωπρόβατα μας λένε πως έχουν σοβαρά προβλήματα γιατί υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Δεν πέφτουν τα ενότια από τα ζώα. Η τεχνολογία δεν λειτουργεί. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε στα βοηδή. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε εθελοντικό και στο μέλλον μέχρι να οριμάσει τεχνολογικά το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να αναπτυχθεί ή να εισαχθεί ποτέ. Αλλά για να τα αφήσουμε να οριμάσει χρειάζεται χρόνος. Και επιπλέον είναι σημαντικό ακριβώς για τη δημόσια υγεία να ε, αμφισβητούμε την ηλεκτρονική σήμανση εάν δεν λειτουργεί. Για τη δημόσια υγεία χρειαζόμαστε 100% σιγουριά. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά, εγώ λέω να μείνουμε στο εθελοντικό σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπάφταν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, έχω σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα των βοηδών. Πολλές φορές έχω καταγγείλει εδώ πέρα την ηλεκτρονική ταυτότητα των προβάτων. Ελπίζω να έμαθε από τα παθήματα της η Κομισιόν στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν ήδη πολλά προβλήματα. Πρέπει, εάν εισαχθεί αυτό το σύστημα, να είναι σε εθελοντική βάση και να μην εξαρτάται το τι θα γίνει από μια έκθεση που θα υποβληθεί σε πέντε χρόνια για την υποχρεωτική χρήση του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα Ταυτοποίηση των βοηδών λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να είναι επιλογή του κάθε αγρότη το να ε, περάσει στο άλλο σύστημα ή όχι, χωρίς τον φόβο της ποινή μέσω της πολλαπλή συμμόρφωση. Επίσης μην ξεχνάμε πως ε, όσον αφορά τα πρόβατα είχαν προβλήματα καθώς ο εξοπλισμός ε, είχε μεγάλες φορές λόγω της έκθεσης στα στοιχεία της φύσης. Το ίδιο είναι αναπόφευκτο και στα βοηδή. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στον τομέα αυτών του Ηνωμένου Βασιλείου και μόλις τώρα ανακάμπτει ο τομέας των βοηδών και βεβαίως πιέζονται και οι δύο τομείς από τις φθηνές εισαγωγές και την αύξηση των ζωοτροφών. Εάν λοιπόν δεν επιτύχει η εισαγωγή αυτού του σήματος από την Κομισιόν θα γονατίσει αυτός ο κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Φερνάντες. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα η ασφάλεια των τροφίμων είναι κάτι που ανησυχεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές. Πρέπει να την εγγυηθούμε, πρέπει να δίδουμε πληροφόρηση πολύ συγκεκριμένη, πολύ σαφή και βάσει μιας πολύ απλής ε, διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ετικετοθεσία του βόλου κρέατος, ώστε να μην δίδονται εσφαλμένες πληροφορίες στον καταναλωτή. Πρέπει να αναφέρεται η ράτσα, ο τρόπος εκτροφής των ζώων, ε, μεταξύ άλλων. Το βόλιο κρέας είναι ένα προϊόν πολύ ευαίσθητο θα έλεγα στην κοινοτική αγορά και υφίσταται τις πιέσεις ανταγωνιστικών προϊόντων αναλόγων από τρίτες χώρες όπου οι απαιτήσει για την καλή διαβίωση των ζώων είναι πολύ χαμηλότερες από τις δικές μας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα της ετικετοθεσίας, να είναι όμως σαφείς, ξεκάθαροι οι κανόνες και το σύστημα ελέγχου να είναι ίδιο για όλα τα κράτη-μέλη ακολουθώντας πάντοτε την κοινοτική λογική. Δηλαδή να μην είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικές δράσεις και τελικά να υπάρχει στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη αυτό το οποίο ήδη ισχύει για τα πουλερικά ε, και για τα αυγά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Τανασέσκο, έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ στο εξή. Παρόλο που η ηλεκτρονική ταυτοποίηση του βόλου κρέατος ίσως είναι επαχθή οικονομικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία ε, για την ε, ασφάλεια των τροφίμων. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι υποχρεωτικός είτε είναι εθελούσιος ο, ο χαρακτήρας της ετικετοθεσίας αυτής, σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη θα πρέπει υποχρεωτικώς να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Θα πρέπει να στηρίξουν είτε με κρατικές ενισχύσεις είτε με υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ανάπτυξη υπαίθρου, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους κτηνοτρόφους. Οφείλουμε να βελτιώσουμε τις βάσεις δεδομένων και να έχουμε καλύτερη ε, αντίδραση όταν θα υπάρξει κάποια αιστεία ε, μολυσματική. Είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους ε, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στη διαχείριση των άμεσων πληρωμών που δίδουμε στους αγρότες. Άλλωστε, βελτιώνεται και η ποιότητα των πληροφοριών που δίδονται στον τι; Εάν τελικά ε, διατηρηθεί η εθελούσια ετικετοθεσία του βοηού κρέατος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπιζότο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η κυρία Μπιζότο, συγγνώμη. Το να καταργηθεί η θεωρητική θυσία του βοηού κρέατο είναι αντιπαραγωγικό και δεν, κάνει, δεν έχει νόημα και για του καταναλωτέ και για του νοοτρόφου στην Ευρώπη. Λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε του καταναλωτέ και να εγγυηθούμε και τη διαφάνεια. Αλλά στην πράξη τελικά ακολουθούμε την αντίθετη κατεύθυνση. Το να μην υπάρχει το σύστημα αντικετοθεσία που εγγυέται πραγματική επίγνωση του τι αγοράζει κανεί. Με αυτή τη διάταξη ευνοείται το ανώνυμο, η παραχάραξη των προϊόντων εις βάρος των κτηνοτρόφων που θέλουν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα. Στην Ιταλία ε, από το εξωτερικό προστέχεται μια μπριζόλα στις δύο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστον από πού προέρχεται. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε την προέλευση, τη ράτσα και τη διατροφή του ζώου. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει αυτό το σύστημα δικαιοθεσία που είναι εντελώ προαιρετικό και λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι πολίτε έχουν ένα καθαγιασμένο δικαίωμα να ξέρουν τι αγοράζουν και τι τρώνε. Αυτό είναι ο δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη. Στην ε, έκθεση που καλούμε θα αναψηφίσουμε αύριο αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Ελίζα, για το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Σοφή Οκονή, η οποία έκανε πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα. Δεν ήταν απλή υπόψη στην Επιτροπή λόγω των διαφορετικών απόψεων και δεν αποτελεί μυστικό όπως και εντός της ομάδας. Είχαμε διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω πως έχουμε τώρα μια καλή βάση για διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο Υπουργών. Για εμά, λοιπόν είναι η πρώτη προτεραιότητα η προστασία των καταναλωτών. Αντλήσαμε τα διδάγματά μα από την κρίση της φωκόδους εγκεφαλοπάθεια. Ταυτόχρονα όμω ξεκαθαρίσαμε στου γεωργού μα πώ θα ελέγξουμε ακόμη περισσότερο τι εισαγωγέ για την τήρηση των κανόνων που έχουμε και δεν θα έχουμε περιττή γραφειοκρατία. Και τώρα θα πρέπει να δούμε που ε, επιτυγχάνουμε τη μέγιστη προστασία των καταναλωτών χωρίς άχρηστη ε, γραφειοκρατία. Οπότε έχουμε εδώ πέρα εμείς ε, μια διευκρίνηση στο άρθρο 1 σημείο 14 που αφορά την ένδειξη των τροφίμων εκείνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εθελοντικό σύστημα. Βεβαίω ο κύριος Νέλχαρτ λέει πώς θα είμαστε σίγουροι πως δεν θα έχουμε εξαπάτηση των καταναλωτών. Μα υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές και οι αναγκαίες κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση βεβαίω. Θα πάμε μετά την ευρυνή ψηφοφορία στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και νομίζω πως όλοι εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι γιατί πρέπει να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο και ίσως στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών να έχουμε και κάποια νέα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πυρίλο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η τροποποίηση του κανονισμού 1760 του 2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηθών και που καταργεί την ε, εθελοντική ετικετοθεσία του βοήου κρέατος ε, έχει μεγάλη σημασία για την ε, προάσπιση της ποιοτικής κτηνοτροφίας και για την προστασία του καταναλωτού μέσω ενημέρωσης και για την ασφάλεια των τροφίμων. Προτείνοντας την κατάργηση της εθελοντικής αντικειτοθεσίας, αποδυναμώνει αυτές τις στοιχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμποδίζοντας τον καταναλωτή να μπορεί να έχει πληροφορίες συμπληρωματικές όπως το φύλλο, η ηλικία ή η διατροφή των ζώων είναι στοιχεία που θεωρώ θεμελιώδη για δύο λόγους. Θα μπορούν να καθοδηγήσουν τον καταναλωτή προς μία αγορά με μεγαλύτερη γνώση και δίνει και προστιθέμενη αξία στο προϊόν αυτή πληροφορία. Επέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύστημα ετικετοθεσίας στο προιον αυτη η πληροφορια επεκρινε η ευρωπαικη επιτροπη το συστημα ετικετοθεσία στο θελοντικο και τα επιχειρήματά της βασίζονται στο μεγάλο διοικητικό άχθος που δεν αντισταθμίζεται από τα πλεονεκτήματα που αποφέρει. Θα ήθελα να ξέρω από ποιας βάσης ε, βασίζονται αυτοί οι ισχυρισμοί, διότι οι πληροφορίες που δόθηκαν από ανεξάρτητος φορείς ε, θεωρούν ότι είναι συγκρατημένο το κόστος αυτό και δικαιολογημένο διότι εγγυάται μια ενημέρωση που είναι προς όφελος και προστατεύει τον καταναλωτή. Για αυτούς τους λόγους δεν συμμερίζομαι τη διαγραφή των άρθρων 16, 17, 18 που είναι κάτι που εμπεριέχεται στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Σάρμπου, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Στη Ρουμανία το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι ενεργό επαγγελματικά στον ε, αγροτικό τομέα. Έχουμε πολλούς μικρούς παραγωγούς και θα πρέπει να επιδείξουμε μεγάλο αίσθημα ευθύνη ως προς το πόσο θα πλήξει ενδεχομένω η νομοθεσία αυτή την κατηγορία παραγωγών. Για αυτούς λοιπόν ε, τους μικρούς κτηνοτρόφους ή παραγωγούς πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουν όλα αυτά τα δυσνόητα και υπερβολικά γραφειοκρατικά κείμενα. Βεβαίως δεν πρέπει να δεχθούμε κανένα συμβιβασμό ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά ούτε θα πρέπει να υιοθετήσουμε μέτρα που θα ε, κάνουν τη δουλειά ενό μικρού κτηνοτρόφου ή παραγωγού να κινδυνεύσει τελικά. Το κόστος δεν θα πρέπει να το αναλαμβάνει ο μικρός παραγωγός. Ιδίω για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα πρέπει να είναι προαιρετική. Θα πρέπει αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία ε, να χαίρει προστασίας και ενίσχυσης, βοήθειας, ειδικότερα ε, πόσο μάλλον αφού είναι αυτοί που εκτρέφουν καλύτερα τα ζώα, τα πιο υγιή και παράγουν τελικά το πιο υγιές κρέας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, ε, Νίκολσον. Κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγή για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι στο τέλος έχουμε κοινή άποψη ότι αυτή η εθελοντική ετικετοθεσία και η ηλεκτρονική αναγνώριση είναι σημαντικά θέματα και τη συγχαίρω για τη δουλειά που έκανε. Ε, υποστηρίζω το να υπάρξει αυτή η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών αλλά επιθελοντικής βάσεως διότι πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ίσως στο μέλλον μπορούμε να το επεξετάσουμε. Τώρα όμως προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε, όχι υποχρεωτικά. Είμαι υπέρ της αρχής ε, της αναγνωρίσεως των κοπαδιών, των ε, βοηδών, μακροπρόθεσμα. Είδαμε προβλήματα που είχαμε όταν ήταν υποχρεωτικό το σύστημα στα πρόβατα. Τεράστια προβλήματα είχαν οι κτηνοτρόφοι που είχαν ε, πρόβατα και στην Ιρλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Και δεν τελειοποιήθηκε. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, περιμένω να έχουμε την τεχνολογία για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε με τους άλλους εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. για 1,5 λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα των βοηθών, εγώ υποστηρίζω μια εθελοντική προσέγγιση ε, για να μην υπάρχει <coughs> ένα διπλό σύστημα διαχείρισης. Στη θεωρία θα μειωθεί το διοικητικό άχθος στους αγρότες και τις αρμόδιες αρχές. Τα κρατημέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να αποφασίσουν το σύστημα το οποίο βολεύει καλύτερα τους ε, αγρότες, ε, τις αγορές και τη, ε, τον κλάδο της επεξεργασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι περισσότεροι αγρότες δεν χρησιμοποιούν τέτοια στήματα και θα ήταν άδικο να το καταστήσουμε το σύστημα υποχρεωτικό, ειδικά αφού δεν υπάρχει απτό όφελο για τον καταναλωτή και φορολογούμενο. Στα δε πρόβατα έχει αποδειχθεί πω είναι μόνο άχρηστη γραφειοκρατία από την Κομισιόν δεν υπάρχει 100% ακρίβεια καθώς η τεχνολογία δεν ε, λειτουργεί και αν δεν ε, επιδείξει ρεαλισμό η Κομισιόν θα τιμωρηθούν αδίκως οι αγρότες στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα των εγωπροβάτων πριν περάσουμε σε άλλους ε, κανόνες για τα βοηδή. Βεβαίω θα μπορούσαμε με την ευελιξία να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι γραφειοκρατικό, θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και θα δίνει στους καταναλωτέ πληροφορίε για να κάνουν τι επιλογέ του. Είναι πράγματι ε, πολλά αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ. Τώρα, μέσω τη διαδικασία Catch the Eye, δίνουμε το λόγο στου αγορητέ. Ε, συνάδελφε Νικολέσκου, έχετε το λόγο. președinte. colegilor care au salutat până acum propunerea Comisiei de Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ανέκαθεν ήμουν υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του βόλιου κρέατος ε, σε προαιρετική βάση. Προφανώς υπάρχουν πλεονεκτήματα ως προς την ιχνηλεσιμότητα. Θα πρέπει να είναι προαιρετική η χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου και θα πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να επιβάλλουν υποχρεωτικό χαρακτήρα χωρίς όμως να ε, θέσουν εν κινδύνο τη δραστηριότητα των μικρών παραγωγών και κτηνοτρόφων. Ο καταναλωτής πρέπει να κάνει ενημερωμένη επιλογή. Το σύστημα πρέπει να είναι σαφές και να μην ε, προσθέτει περαιτέρω επαχθείς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. έχετε λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την συγγήτρια. Βεβαίως, θέλουμε απλοποίηση, μείωση της γραφειοκρατίας και λιγότερα ε, έξοδα και παρόλα αυτά θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Και τρίτον, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η κατάσταση εφαρμογή στα κράτη-μέλη διαφέρει πάρα πολύ. Και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να απαγορεύσουμε την ε, ηλεκτρονική ταυτότητα, αλλά να μην την καταστήσουμε και υποχρεωτική. Γι' αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι εθελοντικό. Γι' αυτό ο συμβιβασμός με βάση ένα εθελοντικό σύστημα είναι ο σωστός. Και πέμπτον, θεωρώ πως θα πρέπει να επανυποβληθεί ο κανονισμός και όχι σε 10 χρόνια. Μην ξεχνάμε πως ε, έχουμε ήδη καεί μία φορά στο χυλό, δηλαδή στην εφαρμογή του σύμματος στα πρόβατα και δεν θέλουμε να πάθουμε το ίδιο πράγμα και στα βοηθή. Ευχαριστώ. Σκότα. Συνάδελφε Σκότα. Αγαπητέ συνάδελφε, σαν πνευματικό μέλο τη Επιτροπή Γεωργία και μέλο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, μάλλον και κανονικό μέλο τη Επιτροπή Γεωργία, είχα δυνατότητα να επεξεργαστώ το θέμα. Από τη μία πλευρά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτό το θέμα δεν λαμβάνει υπόψη τα διάφορα τους διάφορους φορείς, του βασικούς παραγωγούς και του νοτρόφου. Οι προτάσει θέλουν να απογορεύσουν την θελοντική τικετοθεσία είναι ένα μέτρο μη υποχρεωτικό που επιτρέπει στου παραγωγού που επιλέγουν να το κάνουν να δώσουν κάποιε πρόσθετε πληροφορίε στην ετικέτα εφόσον οι ίδιοι εκπροσώποι των κοινοτρόφων ζήτησαν να συνεχίσει να προβλέπεται αυτό το μέτρο, είναι παράδοξο να μην επιτρέπεται αυτή η δυνατότητα. Στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου επεξεργαζόμαστε μέτρα ώστε οι γεωργοί μας να μπορούν με πιο διαφανή τρόπο να μπορούν να κοινοποιούν τα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα που πολλούν φαίνεται να είναι αντιπαραγωγικό. Από την, άλλη πλευρά, από τη μια πλευρά να εργαζόμαστε υπέρ διαφάνεια, ενημέρωση προστασία του καταναλωτού και από την άλλη να απαγορεύουμε μέτρα που ακριβώ εφαρμόζονται θελοντικά και ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Αυτού του είδου η επιλογή γίνεται ε, διότι θέλουμε να μειώσουμε την ποιότητα και τα πρότυπα των προϊόντων των α, γεωργικών. Αλλιώ δεν εξηγείται να πάρω μια παρόν πρόταση. Κατά των γεωργών που θέλουν να αναλάβουν, να δώσουν ποιοτικέ ενδείξει ε, και να διαχωρίζεται το ένα τρόφιμο που ξεχωρίζει από κάποιο άλλο και γι' αυτό το λόγο έχουμε είμαι αντίθετο από αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, Μόλτσερ. Συνάδελφε Μόλτσερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε εφόσον ε, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τα διατροφικά σκάνδαλα που υπάρχουν σε τακτά διαστήματα, καλό είναι το ότι γίνεται μια προσπάθεια αυτή να αποκατασταθεί, αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει με τεράστιο κόστος για τους αγρότες, γιατί ξέρουμε βεβαίως πως το κόστος είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα έσοδα ενός αγρότη, αν σκεφτούμε επίσης το ότι ανεβαίνουν οι ζωοτροφές αλλά ακόμα και το ενίκιο των ε, βοσκοτόπων καθώς ε, υπάρχουν και μέσα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για τους μικρούς αγρότες στην Ευρώπη γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση άντλησε τα σωστά συμπεράσματα εδώ πέρα δηλαδή πως η υποχρεωτική αυτή σήμανση θα έχει μεγάλα οικονομικά μειονεκτήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ, το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, τις διάφορες απόψεις που εξέφρασαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας πω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς πιστεύουμε ότι η πρότασή μας πράγματι θα ωφελήσει τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, αλλά θα βελτιώσει και την ασφάλεια των τροφίμων. Και βεβαίως θα μειώσει το διοικητικό φόρτο ε, για όλο αυτό το κλάδο που έχει να κάνει με το βόλιο κρέας. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κανονισμό ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει ε, το διοικητικό ε, φόρτο ε, και είναι ένας κανονισμός που έτυχε τη στήριξη της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Τώρα, ως προς τα επιμέρους προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ειδική διαδικασία έγκρισης ως εθελούσια ετικετοθεσία για το βόλιο κρέας. Ισχύει η οριζόντια νομοθεσία. Άλλωστε η εθελούσια ετικετοθεσία του βόρειου κρέατος περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και όχι απαραίτητο με την υγεία. Η υγεία και η χνηλασιμότητα ε, είναι πράγματα που εξασφαλίζουμε με, τον, με την υποχρεωτική ετικετοθεσία, όχι με την ε, ετικετοθεσία που γίνεται σε εθελούσια βάση. Για τον λόγο αυτό, κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό ώστε να ξεκινήσει η απαραίτητη διαπραγμάτευση και τελικά να καταλήξουμε ε, στο σύστημα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να το εφαρμόσουμε. Να το εφαρμόσουν όλοι όσοι θέλουν. Και έτσι τελικά ε, θα γίνει λιγότερο ευπαθές το όλο σύστημα και θα μειωθεί και το κόστος ε, για τους μικρούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Δίνουμε το λόγο τώρα στην εισηγήτρια, την κυρία Οκονή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές που εργάστηκαν σε επικοδομητικό πνεύμα. Θα ήθελα σας πω πόσο η δημόσια υγεία για μένα και η υγεία των πολιτών, των ε, πολιτών της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να σας πω ότι επουδενή δεν αμφισβητούμε αυτό το θέμα. Υπάρχει σύστημα αναγνώρισης των βοηδών, ουχή ηλεκτρονικών, αλλά υπάρχει, επιτρέπει, επιτρέπει πολύ ποιοτική ανεχνευσιμότητα. Και δεν αμφισβητούμε αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε να πούμε απλώς αυτό που είπε και ο Σμπάφτον η κυρία Ράιμερς και η κυρία Γκέρλινγκ. Θέλουμε να πούμε ότι η τεχνολογία της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των βοηδών δεν θεωρούμε ότι είναι απόλυτα αξιόπιστη. Περιμένουμε να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι αυτή η αναγνώριση, το σύστημα αναγνώρισης είναι αξιόπιστο για να γίνει υποχρεωτικό το σύστημα. Εξάλλου, εδέχθην ανεφουδεμίας δυσκολίες στις συμβαστικές τροπολογίες να ξαναμελετήσουμε σε μια πενταετία το θέμα, να δούμε αν σημείωσε πρόοδο τεχνολογία, αν επιτρέπει μια καλή ποιότητα ηλεκτρονικής αναγνώρισης, αλλά είναι και πρόβλημα συγκυριακό. Δεν αμφισβητώ και δεν υποβαθμίζω και δεν υπονομεύω την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών λέγοντας ότι θα πρέπει να αφήσουμε ο γεωργικός τομέας του βοήου να έχει χρόνο με φυσικό τρόπο να επιβάλλει αυτή τη νέα τεχνολογία. Αφορά κόστος. Ένα ευρώ αναζώο κοστίζει το ενότιο το ηλεκτρονικό με το τσιπάκι. Θέλουμε μετά σύστημα ανάγνωσης, λογισμικό, που είναι πολύ δαπανηρό. Και οι γεωργοί μας υποφέρουν από την οικονομική συγκυρία και από την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, προς την κυρία Μπιζότο να πω ότι δεν θέλω να καταργηθεί η εθελοντική ετικετοθεσία, όχι. Όπως το είπε πολύ καλά η κυρία Επίτροπος, δεν θέλουμε να καταργήσουμε την εθελοντική ετικετοθεσία, αλλά να την απλουστεύσουμε και σε σύστημα και σαν διαδικασία. Ό,τι αφορά την υγεία των συμπολιτών, αναφέρεται στην υποχρεωτική ετικητοθεσία. Δεν αμφισβητούμε, δεν υπονομεύουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικετοθεσία. Κλείνοντας, υπόθηκε ότι υπάρχει νομικό κενό, το είπε συνάδελφος, όσον αφορά την ετικετοθεσία. Σας λέω όχι. Θα πρέπει να σεβαστούμε τον κανονισμό 1169 κάθετος 2011 όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών. Αυτό που είπατε κύριε Επίτροπε. Είναι η οριζόντια νομοθεσία αυτή που αφορά όλα τα είδη κρεάτων. Το βόλιο κρέας θα είναι στην ε, ίδια βάση όπως όλα τα άλλα είδη κρέατος. Όλες οι τροπολογίες, όλες οι τροπολογίες που κατέθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθετήθηκαν. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους βουλευτές που ακολουθούν τη θέση μου και θα υπερψηφίσουν αύριο. Να διευκρινίσω απλώς ότι πάντα Θέλουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Όλα αυτά θέλουμε να γίνουν σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητήσω αύριο την αναβολή της τελικής ψηφοφορίας για το ψήφισμα. Προτείνω εν συνεχεία να πάμε άμεσα σε τριμερή διάλογο και να επανέλθουμε ακολούθως στην Ολομέλεια για να υποβάλουμε στη ψηφοφορία του Κοινοβουλίου το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Οκονή. Περατώθηκε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τώρα, στην ημερήσια διάταξή μας, έχουμε την έκθεση Φλότ όσον αφορά την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από την CIA σε ευρωπαϊκές χώρες. Δίνω το λόγο στην κυρία Φλότρα, το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτούς τους εννέα μήνες που διήρκησε